τώρα οι δηλώσεις του ενός λεπτού σύμφωνα με το άρθρο 105 του κανονισμού και οι ομιλητές βεβαίως πρέπει να γνωρίζουν πως ο ε, συνήθως είναι περιορισμένος ο χρόνος γιατί έχουμε πολλούς ενδιαφερόμενους. Πρώτα απ' όλα τον λόγο λοιπόν έχει η κυρία Εστέρας Φεραγούτ. Παρακαλώ. Gracias, señora presidenta. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συνθήκη της Λισαβόνας στο άρθρο 3 ασχολείται με την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή καθώς και την αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών. Ως προς τη συνοχή θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτός είναι ένας πρωταρχικός στόχος της Ένωσης. Να επιτρέπει δηλαδή την ανάπτυξη των περιφερειών και να μειώνει τις ανισότητες μεταξύ των διαφόρων ε, περιφερειών της Ένωσης. Αυτό επιδιώκει η συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά στηρίζει και τις απομακρυσμένες περιοχές και τις νησιωτικές. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα των επιδοτήσεων για την ε, Μελίγια και τη Θέουτα. Και τέτοιες επιδοτήσεις είναι άκρος απαραίτητες. Οι περιοχές αυτές εξαρτώνται από τις επιδοτήσεις αυτές και για τις μεταφορές τους και για για διάλους λόγους. Θα πρέπει λοιπόν να εγγυηθούμε αυτού του είδους τις επιδοτήσεις και την ελευθερία καθώς και τις ίσες ευκαιρίες. Καλό λοιπόν το Κοινοβούλιο να στηρίξει την περιφερειακή συνοχή και τα συγκεκριμένα μέτρα. Ε, Ευχαριστώ και τώρα τον λόγο έχει ο κύριος Μύρσκι για ένα λεπτό. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζουμε βέβαια πως είναι κακό να λέει κανείς ψέματα. Όταν βεβαίως ε, κάποιος υπόσχεται κάτι και δεν ε, τηρεί μετά αυτή την υπόσχευση, μιλάμε για απάτη. Πριν από 6 χρόνια λοιπόν κατά τη διάρκεια των μεταξιακών διαπραγματεύσεων η κυβέρνηση της Λετωνίας είχε υποσχεθεί στον Επίτροπο της Διεύρυνσης πώς θα λυθεί το πρόβλημα των μη πολιτών αυτής της χώρας. Εξακολουθεί λοιπόν η Λετωνία να έχει 300.000 κατοίκους οι οποίοι δεν έχουν καθεστώς. Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει μόδα αυτό το πράγμα. Ίσως δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθο αν θεωρώ πω θα πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστώ. Ο Κρι Ντέιβι έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολλέ φορέ έχουμε συζητήσει το πρόβλημα τη Γάζας και του οικονομικού αποκλεισμού του Ισραήλ και της δυστυχίας που προκαλεί. Αλλά δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να αναφέρουμε τα θετικά που συμβαίνουν στη Γάζα. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δύο παιδιά έσπασαν ε, δύο παγκόσμια ρεκόρ, με συγχωρείτε, έσπασαν παγκόσμια ρεκόρ. 700 παιδιά ταυτόχρονα χτυπούσαν ε, μπάλε του μπάσκετ, ενώ ένας παρόμοιος αριθμό πετούσε χαρταετού. Όλα αυτά στις θερινές κατασκηνώσεις όπου έχουν κάτι να κάνουν τα παιδιά στις δύσκολε αυτές συνθήκες. Θα πρέπει ίσω να συγχαρούμε αυτά τα παιδιά για το επίτευγμα αυτό και να υπενθυμίσουμε βεβαίω. Πώ ο μισό πληθυσμό Γάζα είναι ανήλικο κάτω των 18 ετών, δεν έχει ψηφίσει για κανέναν, δεν φταίει τίποτα, θέλουν απλά μια φυσιολογική ζωή και κάποιε ελπίδε για το μέλλον. Και ευχαριστώ την UNRWA, τον οργανισμό του ΟΗΕ και όλου του Παλαιστινίου που συνεργάστηκαν για τι θερινέ αυτέ κατασκηνώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριο Αλφονζή, παρακαλώ. Oui, Madame la Présidente, Κυρία Πρόεδρε, ο διεθνή τύπο μα ενημερώνει για κάτι πολύ ενθαρρυντικό στη χώρα των Βάσκων. Ε, η ΕΤΑ κήρυξε ε, παύση πυρός, ε, κάτι που οδηγεί σε μια ειρηνική κατάσταση. Από ό,τι φαίνεται οι στρατιωτικέ δράσει τη ΕΤΑ σταματούν κάτι που ξεπερνάει αυτό που αναφέρει ο τύπος. Και μάλιστα με διεθνή έλεγχο, όπου θα συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Βόρειο Ιρλανδία η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη συνεισέφερε αποφασιστικά στην κατάκτηση και την εδραίωση της ε, ειρήνης από το 1998 και μετά. Και στη χώρα των Βάσκων θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μεγάλες ευθύνες, γιατί η ελπίδη δεν θα πρέπει να παρεμποδιστεί από τις προκαταλήψεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποφελθεί όλες τις ευκαιρίες που του δίνονται για να προωθήσει την ειρήνη. Κυρία Πρόεδρε, επιμένω και πάλι ότι το βασικό πρόβλημα είναι στην καρδιά της Ευρώπης. Είναι σημαντικό για τη δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεισφέρει δραστήρια στην εδραίωση της ειρήνης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα κύριος Φόξ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, περνούν ε, περίοδο ε, περικοπών και ε, δημοσιονομική δημοσιονομικής πολιτικής. Η, ε, φορολογούμενοι παρόλα αυτά αναγκάζονται να χρηματοδοτήσουν αυξημένε δαπάνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και που αυξάνονται κάθε χρόνο. Οπότε α πρέπει να διαρωτηθούμε, γιατί είναι προτεραιότητα του, Κοινοβουλίου η προστασία των συμφερόντων της, ε, των φορολογουμένων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, δεν θα έπρεπε να μειώνουμε τον προπολογισμό μα, δεν θα έπρεπε δεν είναι παράξενο ε, η δημοσιονομική πειθαρχία να εφαρμόζεται μόνο στις χώρες μέλη, στα κράτη-μέλη και όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, οι αποδοχές παγώνουν και μειώνονται. Ε, δεν θα έπρεπε να δείξουμε αλληλεγγύη. Αφού τα κράτη-μέλη μειώνουν τις δαπάνε κατά 20% σε πραγματικούς ε, όρου τα επόμενα πέντε χρόνια, θα έπρεπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει το ίδιο. Το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να ζητήσει από την Κομισιόν να μειώσει τι δαπάνε τη και να επιστρέψει τα ποσά, τα αντίστοιχα ποσά στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κρίση δανείων στην Ευρωζώνη που οδήγησε τη χώρα μου την Ελλάδα με την προτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει αναδείξει το μεγάλο κοινωνικό και δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της συνθήκης της Λισαβόνας έτσι εκτός από τα κοινωνικά πραξικοπήματα που έχουμε παραδείγματος χάρη στην ελλάδα καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις έχουμε και πολιτικά πραξικοπήματα καθώς η νόμιμη κυβέρνηση της ελλάδας δεν λαμβάνει αποφάσεις διότι όλα αυτά καθορίζονται από το μνημόνιο ευρωπαϊκής ένωσης και Διεθνώς νομισματικό ταμείο το ελληνικό κοινοβούλιο δεν αποφασίζει αν εγκρίνει ή απορρίπτει αυτές τις αποφάσεις και όλα αυτά αποφασίζονται με προεδρικά διατάγματα. όμως κυρία πρόεδρε και κύριοι ε, συνάδελφοι αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι έχουμε πολιτικό πραξικόπημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς ο χρηματοδοτικός μηχανισμός που φτιάχτηκε σύμφωνα με το άρθρο 122 για να δανειοδοτούνται οι χώρες της ευρώπης δεν έχουν ρωτηθεί οι λαοί δεν έχει ρωτηθεί το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. έχουμε λοιπόν μια μετάλλαξη των θεσμών και γι' αυτό σας παρακαλώ κυρία πρόεδρε να θέσετε το ζήτημα και να συζητηθεί το θέμα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 218 των διεθνών συμφωνιών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Μπάφτον. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Ως Ευρωβουλευτής από την Ουαλία με μεγάλη ανησυχία άκουσα τα σχέδια του κυρίου Λεβαντόφσκι να καταργήσει την Βρετανική επιστροφή. Σύμφωνα με τον κύριο Λεβαντόφσκι δεν δικαιολογείται πλέον αυτή η Βρετανική επιστροφή καθώς έχει αλλάξει ο κοινοτικός προπολογισμό και δεν στέκει πλέον αυτή η επιστροφή. Ε, λέτε πως είστε ειλικρινείς κύριε Λεβαντόφσκι. Πείτε μου όμως γιατί ζητούμε να πληρώσει περισσότερο ο Βρετανός ε, φορολογούμενος. Όπως λέτε κι εσείς μιλάμε για 10 δισεκατομμύρια λίρε τα οποία θα συνεισφέρουν οι Βρετανοί φορολογούμενοι για να υποστηρίξουν το ευρώ ω μέρο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου ενώ θα υποστηρίξουν Ελλάδα, Ουγγαρία και Λετωνία και υπολογίζεται πώ θα πληρώσουμε 23 συνολικά δισεκατομμύρια λίρε για να στηρίξουμε το ευρώ. Πόσα παραπάνω θα πρέπει να πληρώσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει από τι εθνικέ κυβερνήσει να μειώσουν τι δημόσιε δαπάνε, ο δικό τη όμω προπολογισμό αυξάνεται ως πότε θα πληρώνουμε το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κερδίζει ο Βρετανικός λαός. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Χάγκετη. Ε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Στην ε, Ουγγαρία έχουμε την 70η επέτειο της ε, δεύτερης αποφάσεως της ε, Βιέννης. Αυτό ήταν πριν από μία εβδομάδα και πήραμε ξανά μία επαρχία ως ε, Ουγγαρία και διορθώθηκε έτσι μία αδικία της συνθήκης των Βερσαλιών. Με την απόφαση αυτή παραδέχτηκε η Ευρώπη πως η συνθήκη του Τριανών ήταν βεβαίω λανθασμένη. Βεβαίω το Ζίγκενμπουργκεν είχε αποχωριστεί από την χώρα μας ε, ξανά μετά τον ε, Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ελπίζουμε όμως να ενωθεί η Ευρώπη πια και να μην υπάρχουν σύνορα και παρακαλώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι ανοιχτό σε επιθυμίες αυτοδιάθεσης ε, αυτών των ανθρώπων. Εγώ πριν από τρεις μήνες προσπάθησα να ανοίξω ένα γραφείο εκεί πέρα στην Σέκελαντ και διακόπτεται ο μιλητής και η πρόεδρος λέει η κυρία Νεντέλσεβα έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να θίξω ε, το ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην επικαιρότητα και έχει να κάνει με την κατάσταση στο Ρωμά. Ε, ελπίζω οι συζητήσει ε, να είναι καρποφόρε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φροντίσει έτσι ώστε να, γίνεται, να εφαρμόζεται κοινοτική νομοθεσία ενώ δεν θα πρέπει να ακολουθήσει αυτή η πολιτική που ακολουθείται σήμερα στη Γαλλία. Κοιτάξτε, σήμερα αυτό που χρειάζονται οι Ρωμά είναι μια πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική και, και μια βιώσιμη λύση για την ενσωμάτωσή του. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα τη πρόσβασή του στην εκπαίδευση, ε, στην παροχή κατάρτιση που να είναι προσαρμοσμένη και να αποτελεί μέρο στρατηγική του 2020, πρόσβαση στι υπηρεσίε υγεία, ε, οικογενειακό προγραμματισμό και κυρίω να βρεθεί λύση ε, στην μόνιμη ένταξη των Ρωμά στην αγορά εργασία αυτό θα διευκολυνθεί με την απορρόφηση των καταλήλων ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν σωστά τα κράτη-μέλη τα κονδύλια. Δεν θα πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία για να ε, αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αυτό διακόπτει πρόεδρο. Ευχαριστώ. Η κυρία Νταντσίλα έχει τώρα τον λόγο. Η Σέγγεν είναι ένας ε, κοινό χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας και νομίζω ότι η Ρουμανία πληρεί τα απαραίτητα κριτήρια ε, δεδομένου ότι έχουν γίνει και οι κατάλληλες αξιολογήσεις. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από όλες τις αποστολές αξιολόγησης της Ρουμανίας μέχρι τώρα και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους. Είμαι επεπισμένη ότι η Ρουμανία μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις ε, μεταναστευτικές ροές από χώρες εκτός Σέγγεν, σεβόμενοι τις προδιαγραφές ε, που έχουν οριστεί για όλες τις χώρες του, του Σέγγεν. Ε, αυτό δεν έχει σχέση με την κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Η νομοθεσία θα πρέπει να έχει ως στόχο να βελτιώσει την κατάσταση των Ρώμα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και να μην, επι... να περικόψει τα δικαιώματά τους θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στην συμμετοχή στι Έγκες Ρουμανία και τη κατάσταση των Ρώμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπιλμπά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καταδικάσω τη στάση του, ε, της κυβέρνησης του Μαρόκο στις 28 Αυγούστου ε, κατά ε, των κατοίκων του Σαχράου. Ε, ε, κοιτάξτε, ε, μιλάμε για παραβίαση των δικαιωμάτων, μιλάμε για την Κούβα, για την Ονδούρα, όμω αυτή τη φορά δεν το πράξαμε και εδώ διακυβεύεται η εξεπιστία μα και, και, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και επειδή μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα και ω Ευρωπαία και ω προερχόμενοι από τη χώρα των Βάσκων, η χθεσινή κατάπαυση του πυρό δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Θέλουμε να είναι οριστική και να μπορεί να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητα τρίτα μέρη θέλουμε να καταδικάσουμε για πάντα και να παρνηθούμε για πάντα ε, τη βία. Το μέλλον τη χώρα των Βάσκων βρίσκεται στην κοινωνία των πολιτών τη χώρα αυτή, τη περιοχή αυτή ε, και στου ε, εκλεγμένου με δημοκρατικό τρόπο. θα καταβάλω κάθε προσπάθεια έτσι ώστε ε, να υπάρξει επίλυση του προβλήματο αυτού. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ο επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Μιγκάλσκι pani przewodnicząca! kiedy byliśmy na wakacjach niestety u naszego partnera wschodniego czyli. στην ε, ρωσία γίνονται καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, αυτές οι καταπατήσεις είναι συνεχείς στην Κουσιατία και τον Ταγκιστάν γίνονται απαγωγές ε, δεν επιτράπηκαν διαδηλώσεις 31 Αυγούστου όπως επίσης και την 1η Σεπτεμβρίου και τις 30 Αυγούστου. Έγιναν συλλήψεις ε, αντικαθεστωτικών, ε, γνωστά ονόματα, κατά τη διάρκεια μια συναυλία στην ε, Μόσχα, ε, η, η διεθνής, ε, το γραφείο της Διεθνούς Αμνηστίας κατασχέθηκε και καταστράφηκε δυσάρεστες ιστορίες όλοι θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας όταν συνομιλούμε με τους ανατολικούς εταίρους μας. Ευχαριστώ κυρία Φιγκερέδο. Ε, Αυτό το καλοκαίρι ούτε και η εποχική εργασία μείωσε ε, την ανεργία σε ποσοστό κάτω από 10%. Έχει φτάσει σε πάνω από 20% μεταξύ των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Eurostat η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και οι κυβερνήσεις δεν δίνουν όμως προτεραιότητα σε αυτό το πρόβλημα. Ε, επιμένουν στην αυστηρή τήρηση του συμφώνου της, ε, του Μάστριχτ ε, και με αυτόν τον τρόπο καταδικάζουν την, την, τους νέους μας ε, κάτι που συνοδεύεται μάλιστα και με ε, εκδίωξη και επιστροφή στη χώρα τους μεγάλων ομάδων όπως τον Ρωμά. Ε, πρόκειται για φαινόμενα απαράδεκτα, ρατσιστικά, ξενοφοβικά που καθιστούν σαφές ότι η ελευθερία της κυκλοφορίας αφορά μόνο τα αγαθά και τα κεφάλαια και το κεφάλαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προασπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερνάντεθ κατόπιν. Δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κάθε χρόνο καίγονται εκατοντάδες χιλιάδες εκτάρια από πυρκαγιές. Στην ε, Πορτογαλία κάηκαν πάνω από 100.000 εκτάρια φέτος. Και σε προστατευμένες περιοχές ε, δεν διαφεύγουν του κινδύνου. 8.000 εκτάρια κάηκαν από προστατευμένε περιοχέ φέτο στην Πορτογαλία. Καταστρέφεται έτσι η πολιτική μα και η ψυχή μα ε, κληρονομιά ε, και πλήττεται θανάσιμα η βιοπικιλότητα, καταστρέφονται υποδομές και χειροτερεύουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επενδύει στην πρόληψη των πυρκαγιών. Από την άλλη μεριά, πολλές από αυτές τις πυρκαγιές είναι ε, αποτέλεσμα της απερίμωσης και των, της έλλειψης πολιτικών για την ε, Ήπεθρο. Είναι κρίμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναλαμβάνει ε, εκστρατεία πρόληψης ε, των πυρκαγιών με ενίσχυση των προγραμμάτων υπέρ της Ήπεθρου. Ευχαριστώ κυρία Κρετού. Se împlinesc trei luni de când uh, printre vicepreședințele uh, Parlamentului European se numără domnul. Ευχαριστώ. Τρεις μήνες uh, πέρασαν μετά από την εκλογή του αντιπροέδρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από αμφιλεγόμενες εκλογές και ορισμένοι ε, επιστήσαμε την προσοχή ε, ε, στο ζήτημα της εκλογής κάποιου που προωθεί ε, αποσχιστικές τάσεις και κυρίως ε, αν λάβουμε υπόψη τις προσπάθειες των νέων κρατών μελών για να ξεπεράσουν τα, προτάσεις τα σφάλματα του παρελθόντο. Δυστυχώ όμω ο κύριο Τόκια ε, προωθεί ε, τα σοβινιστικά και εξτρεμιστικά μηνύματα. Ε, καλή για την επίτευξη τη απόσχηση ορισμένων περιοχών τη Ρουμανία. Μιλάμε δηλαδή για κάποιον ο οποίο καταφέρεται ει βάρο τη εδαφική ακαιρεότητα μια συγκεκριμένη χώρα. Δεδομένη τη τάση του, ζητώ να παραιτηθεί από το αξίωμά του. Ευχαριστώ κύριο Τρεμόσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπω ε, ξέρετε, την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώσαμε τι διαπραγματεύσει για το πακέτο κρηματοοικονομική επιτήρηση που θα ψηφιστεί στην επόμενη Ολομέλεια. Μέχρι τέλους ε, υποστηρίξαμε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να γίνει ε, αυτόματα για τα πέντε πρώτα χρόνια ο πρόεδρος, να γίνει πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκού Συστημικού ε, Κινδύνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, θα συμμετάσχει πολύ περισσότερο στην χρηματοοικονομική επιτήρηση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών, χρηματοοικονομικών αγορών και οργάνων. Αυτό σημαίνει επίση ότι ο κ. Τρισέ στι τακτικέ ακροάσει του εδώ πέρα θα χρειάζεται να απαντάει σε ερωτήσει και σχετικέ με την χρηματοοικονομική πολιτική και όχι μόνο σε σχέση με τη σταθερότητα των τιμών. Ω φιλελεύθερο, πιστεύω πιο πολύ στι μεταρρυθμίσει παρά σε επαναστάσεις. Ε, χάρη σε αυτή τη μεταρρύθμιση, ε, θα είναι πολύ πιο δύσκολο τα χρηματοπιστωτικά ε, όργανα να συνεχίσουν να δημιουργούν κρίσει όπω αυτή τελευταία. Ευχαριστώ, η κυρία Μαρίσα Ματιάς. Πριν από μερικά μέρες σε μια ε, επιχείρηση υποδημάτων ε, ε, εκδιώθηκαν και έχασαν τη δουλειά τους όλες οι ε, ε, υπάλληλοι μιας βιομηχανικής εξαιτίας ενός απλού μηνύματος SMS. είναι φανερό το ότι εξακολουθούν να παραβιάζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή έχουμε, πάνω, έχουμε 8 εκατομμύρια καινούριου ανέργου σε ένα σύνολο 25 εκατομμυρίων. Και εξακολουθούμε να βλέπουμε τέτοια ε, επεισόδια που ντροπιάζουν την παράδοσή μα. Έχουμε μια παράδοση προστασία των, των δικαιωμάτων των ε, εργαζομένων. Χρειάζονται περισσότερα μέτρα όμως και θα πρέπει να πάρει μέτρα η Κομισιόν. Ποια είναι αυτά τα μέτρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τέτοιου είδους ε, ε, επεισόδια μαζικών ε, απολύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Higgins. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Anglo-Irish Bank φαίνεται πως έγινε συνώνυμη των απερισκεψιών της, ε, του τραπεζικού τρομέα. Μα είχαν πει πω οι διάσει χρειαζόταν 25 δισεκατομμύρια ευρώ, τώρα τελικά είναι 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά είναι εικασίε. Η κυβέρνηση δεν γνωρίζει το ποσό. Μιλάμε όμω για 210 εκατομμύρια ευρώ την εβδομάδα. Και 8,2 δισεκατομμύρια ήταν οι ζημίε του πρώτου εξαμήνου και η κατάσταση χειροτερεύει. Ο Υπουργό Οικονομικών τη Ιρλανδία είναι στι Βρυξέλλε αυτήν την εβδομάδα και ζητάει έδεια να συνεχιστεί η διάσωση. Εγώ ζητάω από την Κομισιόν και την Επίτροπο Ανταγωνισμού να του πούνε ομά ότι πρέπει να κλείσει η τράπεζα όχι σε 10 χρόνια όπω θέλει η κυβέρνηση αλλά σε 2 ή 3 χρόνια. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Ευχαριστώ. Κυρία Μουνιέση, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή στην Χιλή 33 ε, ανθρακορίχοι βρίσκονται κάτω ε, από το έδαφος και περιμένουν τη διάσωσή, του. τους. Ε, έχουν την υποστήριξή μας και την υποστήριξη όλων των σοσιαλιστών της Ευρώπης. Αυτοί που υπάρχουν στην Αστούρια, στην Αραγόν, στη Βαλένθια που βρίσκονται στα, στα, στα, στα πηγάδια αυτή τη στιγμή σε αυτές τις περιοχές όλοι αυτοί οι ανθρακορίχοι. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση τοποθετείται για το βασιλικό διάταγμα της Ισπανίας ε, και για την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και στην ουσία ε, θα αποφασίσει ε, για, την, για το μέλλον 44.000 οικογενειών στην Ισπανία. Το ζήτημα είναι κατά πόσον θα υπάρξει, θα επένδυση σε σύγχρονη τεχνολογία. Από αυτό εξαρτάται η ζωή πολλών περιοχών της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Αστούριας. Εδώ μιλάμε για μια αυτόχθονη μορφή ενέργειας. Πρέπει να καταλάβει το πόσο μεγάλη σημασία ε, θα έχει η απόφαση της, ε, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και για ολόκληρο το μέλλον του τομέα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριος Χάγκλουντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πέρσι η Επιτροπή Αλληλείας του Κοινοβουλία μας καταψήφισε την ανανέωση της Συμφωνίας Αλληλείας με την Γουινέα Κονάκρη μετά από μια σφαγή που είχε γίνει εκεί. Το τον Αύγουστο προετοιμάζονταν οι εκλογές, ε, οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές από το 1958. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποστείλει και παρατηρητές σε εκλογές αυτές και θα παρακολουθούμε την κατάσταση ε, έτσι ώστε οι εκλογές αυτές να είναι δημοκρατικές. Το κομμάτι και του κόσμου είναι ένα μέρος στο οποίο πρέπει να βοηθήσουμε να έρθει προς την δημοκρατία. Όλη η περιοχή και η Γουινέα Μπισάου είναι προβληματική. Οι εκλογές στην Γουινέα Κονάκρη ήταν τόσο προβληματικές έτσι ώστε είχαμε πολλές αναβολές μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου τελικά λόγω της εκτεταμένης νοθείας. Πρέπει να το σημειώσει λοιπόν αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προσπαθήσει να βελτιώσει την κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κατόπιν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω για το δημοψήφισμα στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Οι πολίτες τοποθετήθηκαν ε, για, την, ε, για τις άμεσες εκλογές ε, του, του Προέδρου που θα οδηγήσει σε απεμπλοκή ε, της ε, ε, πολιτικής κατάσταση. Οι, οι κομμουνιστές ζήτησαν να υπάρξει μποϊκοτάρισμα του δημοψηφίσματος και αυτή η τακτική απέδωσε, δεν υπήρξε αρκετή συμμετοχή στο δημοψήφισμα. Ο συνασπισμό των δημοκρατικών κομμάτων ε, ε τώρα ε, θα πρέπει να ξεπεράσει αυτή την αποτυχία. Θα πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αφήνοντας κατά μέρο την δική μας υπερηφάνεια για να δούμε το πώς η χώρα αυτή θα προχωρήσει προς την κατεύθυνση δημοκρατικής οδού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ κύριο Σίβαν. ναι, κύριε συνάδελφε. Ναι, ναι, εσείς έχετε τον λόγο. Ιβαν Καταλίν. Ε, ναι, εντάξει. Η δημοκρατία της Μολδαβίας ε, βρίσκεται σε ένα δημοκρατικό αδιέξοδο και πάνω από ένα χρόνο. Παρόλα αυτά, η χώρα αυτή έχει κάνει σημαντική πρόοδο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση το χτεσινό δημοψήφισμα θα μπορούσε να βγάλει την Μολδαβία από αυτό το δημοκρατικό αδιέξοδο και να τη φέρει ακόμα πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν κατέστη δυνατό. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί νίκη των κομμουνιστών έναντι του συνασπισμού που είχε ταχθεί υπέρ της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αποτελεί απλώς ένα εμπόδιο στην ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας. Θα πρέπει να την υποστηρίξουμε θα πρέπει να συνεχίσουμε να την ενθαρρύνουμε γιατί έχει αποδείξει πως έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Ευχαριστώ κύριος Κάζακ. Κύριε Πρόεδρε, η οι διαμαρτυρίες ε, ε, των μουσουλμάνων στη Βουλγαρία εντείνονται. Το περασμένο Σάββατο ε, υπήρξε πολιορτία της έδρας του Μεγάλου Μουφτή λόγω της απόφασης ε, τη απόφαση η οποία δεν άφηνε του υπαλλήλου να περάσουν μέχρι το κτίριο αυτό. Λοιπόν, ε, συγκέντρωσαν 230.000 υπογραφές, ε, συγκεντρώθηκαν λοιπόν 230.000 υπογραφές ε, και τελικά υπάρχει μια παράλογη κατάσταση και, και όλα αυτά δείχνουν την παράλογη και την δικτατορική παρέμβαση του, των δικαστικών αρχών στην, στις, στις θρησκευτικέ μειονότητες με βάση την αρχή διέρη και βασίλευε. Ζητώ να υπάρξει ε, συγκεκριμένη εξακρίβωση των γεγονότων εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Επειδή ήρθε τελικά ο κύριο Σίρεν Χάουζερ, έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγα λόγια θα ήθελα να πω για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, παρουσίασα ένα σχετικό εγχειρίδιο σήμερα στην Βιέννη και από την ανάλυση αυτή προκύπτει πως ε, θα έχουμε του χρόνου γύρω στις 40 τέτοιες εκτελεστικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Και αν βάλουμε και αυτές του Συμβουλίου μέσα μιλάμε για 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε έτος και 7.000 άτομα που σε αυτή τη μυστική δεύτερη ευρωπαϊκή γραφειοκρατία. Νομίζω πως η άναρχη αυτή ανάπτυξη απαιτεί να μπουν όλα αυτά τα πράγματα επιτάπητος και να δοθούν λύσεις. Και εγώ έχω ένα πρόγραμμα 11 σημείων για το πώς ετησίως θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε 500 εκατομμύρια ευρώ από τα λεφτά των φορολογουμένων. Όλα αυτά είναι στο site μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νικολάζεκ. Ε, ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το τραγικό γεγονός ε, της προηγούμενης Δευτέρας στην Μπρατισλάβα κόστισε τη ζωή σε 8 άτομα. Συγκλώνησε ολόκληρη την Σλοβακία ένας άνθρωπος σε κατάσταση αμόκ προκάλεσε επίσης πέρα από τους νεκρούς και 15 τραυματίες και τους 8 νεκρούς όπως είπα. Πιθανώς πρόκειτο για ένα άτομο πνευματικά σταθές. Αλλά ε, βεβαίω ε, δεν ξέρουμε εάν ήταν ρατσιστικό το κίνητρο, μάλλον δεν ήταν. Η χρήση ε, δε μιας ειδικής μονάδας απαιτήθηκε για να σταματήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Και βεβαίως ε, υποστηρίζουμε όλα αυτά τα βήματα για τη μεγαλύτερη ασφάλεια του πληθυσμού. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στις επικίνδυνες αυτές ζώνες. Θα ήθελα να προσθέσω πως η Σλοβακική Δημοκρατία ε, θλίβεται πάρα πολύ από αυτά Ευχαριστώ. Yeah, uh, thank you, uh, uh, President. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω τον ρόλο τον οποίο μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την οικονομική ανάκαμψη. Έχει πάρα πολλά κονδύλια στη διάθεσή της. Το πρόγραμμα πλαίσιο 7, τα κονδύλια της αγροτικής πολιτικής και τα διαρθρωτικά ταμεία. Πρόσφατο παράδειγμα καλής χρήσης είναι η ανακοίνωση σήμερα 107 εκατομμυρίων λιρών ε, που θα πάνε σε έργα στην Ουαλία και βεβαίως πάνω από 50% αυτής της χρηματοδότησης προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αναζυγονίσουν τον τομέα αυτόν και θα ήθελα βεβαίως να συγχαρώ και την Ουαλική Συνέλευση και την τοπική κυβέρνηση και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η χρηματοδότηση και το 2011 και στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2013. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κέλλη έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής του 2020 και μάλιστα δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να πτύχουμε χωρίς αυτήν οποιοδήποτε στόχο. Βεβαίως οι χώρες θα προσπαθήσουν να πετύχουν το στόχο των ανανεώσιμων αλλά και αν το κάνουν αυτό θα εξακολουθήσουμε να εξαρτώμεθα από τρίτες χώρες. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες χώρες έχουν διμερείς συμφωνίες, πρέπει να αποκτήσουμε πολυμερείς συμφωνίες σύμφωνα με το άρθρο 194 της Συνθήκης Λισαβόνας και ελπίζω να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα, όπως έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική και πολιτική αλληλείας να φτάσουμε και σε μια κοινή ενεργειακή πολιτική, ειδικά όσον αφορά τις τρίτες χώρες. Για να έχουμε πρώτα απ' όλα ασφάλεια στι ε, προμηθειέ μας και βεβαίως δεύτερον για να μην εκμεταλλεύονται τις διαφορέ χώρε όπως η Ρωσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Σάμπου έχει κατόπιν το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, η διατροφή έχει να κάνει με την ε, σωματική και την ψυχική εξέλιξη του ανθρώπου. Ε, μία μη ε, υγιής διατροφή μπορεί να οδηγήσει σε διαβήτη, σε καρκίνο, σε καρδιακά νοσήματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρξει η σωστή ενημέρωση τόσο των ενηλίκων αλλά και κυρίως των παιδιών. Τα σχολεία θα μπορούσαν να παίξουν εδώ ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να προωθήσουν την υγιή διατροφή. Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα ανισχυτικό γεγονός. Στις βλαβερές συνέπειες ε, το που έχει ε, το fast food. Θα, ε, νομίζω λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπα-Νικολάου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε όλοι μας τονίζουμε την ανάγκη για επένδυση στην παιδεία στην κοινωνία της γνώσης και αυτό το κάνουμε με κάθε τρόπο. πρέπει όμως παράλληλα να καταθέτουμε και να καταδικάζουμε τα κακό κείμενα που παρατηρούμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. αναφέρω ένα παράδειγμα στην ελλάδα. στην ελλάδα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εισάγεται ένας μαθητής μετά από εξετάσεις. θεσπίστηκε το προηγούμενο διάστημα από την ελληνική κυβέρνηση το μέτρο της βάσης του 10. Ο μαθητής δηλαδή να πρέπει να γράψει 10 στα 20 προκειμένου να μπορεί να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ελληνική κυβέρνηση πρόσφατα κατήργησε αυτό το μέτρο για λόγους ακατανόητους. Αποτέλεσμα, μαθητής εισήχθη σε σχολή της, τριτο... της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό 0,91 στα 20 αν μη τι άλλο αυτό πρέπει να αλλάξει αν μη τι άλλο όλοι μας πρέπει να καταδικάζουμε τέτοια φαινόμενα προκειμένου να προαχθεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλη την ευρώπη. σας ευχαριστώ πολύ για τον λόγο. Έχουμε μια θετική είδηση, το ότι δηλαδή βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση και στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι οικονομικές προοπτικές της Ουγγαρίας βελτιώθηκαν. Αλλά βεβαίως ε, η διεθνής αξιολόγηση της Ουγγαρίας επιδεινώθηκε και βλέπουμε εδώ πέρα ότι δεν ε, μπορούμε να έχουμε μία μείωση των επιτοκίων και αυτό σημαίνει βεβαίως ε, πως ε, θα χειροτερέψουν τα πράγματα για τους Ουγγρούς πολίτες. Άνθρωποι θα χάσουν τα σπίτια τους. Σας παρακαλώ λοιπόν να βοηθήσετε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην Ουγγαρία και να αλλάξει η αξιολόγηση των διεθνών επενδυτών. Αυτό αφορά βεβαίως πάρα πολλά εκατομμυρία ανθρώπους. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρίγνερ. Ευχαριστώ. Η Μακαρένα δεν είναι μόνο ένας χορός, αλλά και μία μικρή πόλη της Κολομβίας. Το 2009 διαμαρτυρήθηκαν εκεί πέρα οι αγρότες για το δηλητηριασμένο νερό και φαίνεται πως ε, βρέθηκαν σε τάφους 2.000 ανώνυμα πτώματα. Υπάρχει μια οργάνωση που λέγεται Justice for Colombia που ασχολείται ακριβώς με την υπόθεση της ε, Μακαρένα. Πάρα πολλοί άνθρωποι περπάτησαν μέρες μέσα στη ζούγκλα για να μπορέσουν να διηγηθούν τις προσωπικές ιστορίες των αγαπημένων τους που εξαφανίστηκαν και τραυματίστηκαν κτλ. Το αποτέλεσμα ήταν βέβαιως απειλές θανάτου. Είδαμε το μαζικό τάφο και υπάρχει υποψία πως ο ίδιος ο στρατός συμμετείχε στις εκτελέσεις. Δεν υπάρχει καμία χώρα παγκοσμίω όπου εξαφανίζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι όσοι στην ε, Κολομβία. Και μιλάμε για μια ατιμορρησία που φτάνει το 90%. Το να κλείσουμε και συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Κολομβία είναι επιβράβευση αυτής της συμπεριφοράς. Ευχαριστώ. Τελευταίος τον λόγο, τον λόγο έχει η κυρία Γκυγιόν. Θα ήθελα να επιμείνω και πάλι στην κατάσταση του Αμαντίας Τσάνι που έχει καταδικαστεί σε θάνατο και ε, σύντομα θα λιθοβοληθεί. Ε, στην, ε, στην, σε μια βρετανική εφημερίδα δημοσιεύτηκε μια δίθεν φωτογραφία της και καταδικάστηκε σε 99 βροντουλιές επιπλέον δεν ήταν δική της φωτογραφία βέβαια παρόλα αυτά δεν άλλαξε τίποτα ποια χώρα τον 21ο αιώνα έχει στον ποινικό τη κώδικα το μέγεθο ε, τη πέτρα που θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε τέτοιους λιθοβολισμού. Η πολιτική δεν έχει καταφέρει να απομακρύνει, το, να εξαφανίσει το φαινόμενο του λιθοβολισμού. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ως πολίτες για να αποφύγουμε και να, αυτά το φαινόμενο και να σώσουμε τη συγκεκριμένη κοπέλα. Ευχαριστώ. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η έκθεση του κυρίου Πόρτας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Τον λόγο έχει ο εισηγητής για τέσσερα λεπτά. Obrigado,